Έχει τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθεί. Αρχής γενομένης από την αυριανή ημέρα 27 Οκτωβρίου 2017. Ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση μείζων σημασία επερωτήσεων άρθρο 130 β του κανονισμού. Η σημερινή συζήτηση αφορά τι συντονισμένε προσπάθειε Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού.